Ωραία, συνάδελφοι. Ζητούμε και συγγνώμη από τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τα προβλήματα που είχε να έρθει στο κτίριό μα. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Και θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία στο μέλλον. Να σας πενθυμίσω ότι έχουμε αλλάξει την μερική διάταξη. Έχουμε ακυρώσει το σημείο 15 για την γνωμοδότηση για την Επιτροπή Γυναικών για την ε, ισότητα ε, μεταξύ των φύλων στην κλινική έρευνα και το έχουμε αντικαταστήσει με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι πάμε σπίτια μας το βράδυ, βλέπουμε στη τηλεόραση τι συμβαίνει εκεί, τα, τα αποτρόπια αυτά εγκλήματα και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χαλέπι. Έχω μιλήσει με τον Επίτροπο στη Στυλιανίδη και ξέρω ότι και εκείνο και η κυρία Μογκερίνη κάνουν ό,τι μπορούν για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον κόσμο, στο Ανατολικό Χαλέπι. Όμω ε, ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση και σήμερα το πρωί ακούσαμε ότι έχουν στοχευθεί νοσοκομεία. Όπως και στις ε, 19 Σεπτεμβρίου όπου ένα ε, κομβόι δέχθηκε επίθεση και σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι καθώς προσπαθούσαν ε, να διαβιβάσουν βοήθεια προς το Χαλέπι. Ο κύριος Διπουργέ έχει έρθει εδώ λοιπόν, είναι ε, διευθυντής του τμήματος για την Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Θα μας ενημερώσει για τα τι συμβαίνει στην περιοχή αλλά θα μιλήσει και για την IT. Γιατί ξέρουμε ότι και εκεί ε, είχαμε τεράστιες απώλειες ανθρωπίνων ζώων λόγω του τυφώνα το Σαββατοκυριακό. Παρακαλώ όποιος ε, θέλει τα πηγαδάκια να συνεχιστούν εκτός της αίθουσας. Παρακαλώ κύριος Δεμπογιέφ, έχετε λόγο. Εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είχα λάβει υπόψη, δεν είχα υπολογίσει ε, τον χρόνο. Και συγγνώμη που καθυστέρησα. Και μια συνάδελφός μου πρέπει να έρθει για να μιλήσει για την IT. Τα επόμενα λεπτά νομίζω θα είναι εδώ. Ξέρω ότι είναι κάπου μέσα στο κτίριο. Τα είπατε όλα, κυρία Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα και να ζητήσω συγγνώμη, αλλά και να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή σα για τον τρόπο με τον οποίο και εσεί παρακολουθείτε αυτέ τι εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις και για τη στήριξη που μας παρέχεται και με την συζήτηση στην Ολομέλεια και με το ψήφισμα κατόπιν της ε, συζήτησης στην Ολομέλεια. Ήταν ε, πολύ σημαντικές κινήσεις για εμάς και έχουμε πραγματικά την εντύπωση ότι προσπαθώντας κι εμείς να συνεισφέρουμε όχι στη λύση, δεν την αποκαλύψω λύση προβλήματος, αλλά τουλάχιστον στο να υπάρξει κάποια πρόοδος ή να περιορίσουμε την ε, περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής ε, κατάστασης. Προσπαθούμε αυτή την πολιτική στήριξη μας παρέχεται να τη μεταφράσουμε σε έργα. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Επίτροπος Τηλιανίδης μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο Αντιπρόεδρο Μογκερίνη πριν από 10 ημέρες είναι γνωστή σε εσάς Μέχρι τότε διαδραματίσαμε και εμείς το ρόλο μας ε, στην ε, Task Force στην ανθρωπιστική. Ε, τμήμα της διαδικασίας της οποίας ηγήθηκε ο Στέφαν Μιστούρα στην Γενέβη. Ξέρω ότι είχαμε δύο task force, αυτή, η ανθρωπιστική και η task force για την εκεχηρία. Προσπαθήσαμε κατά το δυνατόν να ε, στηρίξουμε τις προσπάθειες ε, όλων όσοι ήθελαν να διευκολύνουν την πρόσβαση για ένα διάστημα. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Υπήρχε αποτέλεσμα αυτών, αυτής της ανθρωπιστικής task force. Υπήρξε αυτή η συνένεση σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση ενός ε, μηχανισμού οικοδόμησης εμπιστοσύνης και νομίζω ότι βοήθησε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες ε, απομακρυσμένες ε, δυσπρόσιτες περιοχές και μετά όλη η δικασία και πάλι πολιτικοποιήθηκε. Τα ξέρετε κι εσείς αυτά με την πολιτική ζημία και άλλα ζητήματα και έτσι κολλήσαμε. Παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι βέβαια η προσοχή όλου του κόσμου έχει στραφεί στο Ανατολικό Χαλέπι. Όμω αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι πολύ δραματική η κατάσταση βέβαια, αλλά το παγόβουνο αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε λοιπόν στο Χαλέπι είναι απλώς μία συμβολική κίνηση, μια, συμβολική συζήτηση, μια δοκιμή ε, για το θερπιστικό ζήτημα, το οποίο ελπίζουμε να μας οδηγήσει στην εξέβρεση μια ε, λύση ω προ την πρόσβαση και ω προ την εκένωση. Όμως ε, είναι πραγματικά το δέντρο και όχι το δάσο, Γιατί το δάσο τη ανθρωπιστική ε, καταστροφή στην Συρία γίνεται κάθε μέρα όλο και μεγαλύτερο. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω επίση ότι πρέπει να έχουμε μια συνολική αντίληψη τη κατάσταση, Ξέρουμε ε, τι μαγειρεύεται αυτή τη στιγμή και στη Μοσούλη στο Ιράκ. Πολύ φοβάμαι ότι θα έρθει η στιγμή και δεν απέχουμε και πολύ από εκεί που θα έχουμε ταυτόχρονα και Χαλέπι και Μοσούλη, ενδεχομένως και Ράκα. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς ε, θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και εδώ δεν αναφέρομαι στις γεωπολιτικές ε, επιπτώσεις των όσων θα μπορούσαν να συμβούν εκεί. Απλώς περιορίζομαι μόνο στο πώς θα καταφέρουμε να καθοδηγήσουμε αυτή την ανθρωπιστική διαδικασία. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που, που θέλουμε να αποστείλουμε. σε όλε αυτές τις εκκλήσει που απευθύνθηκαν από τον Επίτροπο Στυλιανίδη και από την ε, Αντιπρόεδρο Μογκερίνη. Εδώ και δέκα ημέρες με πολύ ενεργό και δραστήριο τρόπο προωθούν αυτό το μήνυμα. Είναι λοιπόν μια ανθρωπιστική διαδικασία και επιχείρηση. Τάχιστα επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κατάσταση και πρέπει να επανέλθουμε στις βασικές αρχές της ε, ανθρωπιστικής παρέμβασης και κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν ε, επιτρέπεται ε, να καταλύεται αυτή η αρχή για λόγους πολιτικούς. Ξέρουμε ότι έχουμε δύο δράσεις υπό την ίδια ομπρέλα, η ιατρική εκένωση Και δεύτερον, η παροχή βασικών, βασικού εξοπλισμού και άλλων βοηθημάτων ε, νερού, τροφής στον ε, τοπικό πληθυσμό. Όλοι οι εταίροι είναι έτοιμοι. και ο ΠΟΗ και ο Ερυθρός Σταυρός, βασικός μας εταίρος σε αυτή την επιχείρηση. Εμείς έχουμε δώσει μία ε, γραμμή πίστοσης 25 εκατομμυρίων ευρώ που είχε προβλεφθεί στον προπολογισμό μας για να αντλήσουμε από εκεί κονδύλια και να στηρίξουμε οποιαδήποτε ε, επιπλέον παρέμβαση. Μαζί με τα κράτη-μέλη εξετάζουμε τη δυνατότητα να συστήσουμε και μία δεύτερη γραμμή ιατρικής εκένωσης, δηλαδή εάν υπάρξει εκένωση σε ένα από τα τρία ε, σημεία που ήδη προβλέπονται για αυτούς, αλλά δεν, δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι και έτσι δεν λαμβάνουν την ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται, ενδέχεται να μπορούμε να τους φέρουμε σε ένα ευρωπαϊκό νοσοκομείο. Όλα αυτά τα εξετάζουμε και τα τελειοποιούμε κάθε μέρα, όμως, βέβαια, χρειαζόμαστε αδειοδότηση για να έχουμε, για να έχουμε είσοδο, πρόσβαση, έξοδο. Υπό κανένα χρονικό περιορισμό. Είναι εξαιρετικά λεπτή η επιχείρηση αυτή και όταν έχουμε 48 ώρες πριν αρχίσουν και πάλι οι μοβαρδισμοί, όπως ήταν η συμφωνία που είχε προταθεί προηγουμένω, αυτό δεν δουλεύει. Είναι ανθρωπιστική επιχείρηση που θα πρέπει να εφαρμόζεται ε, υπό ελάχιστες προποθέσει τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει με του εταίρου μα και ευρύτερα με την ε, Συριακή Κυβέρνηση για να λάβουμε αυτές τις αδειοδοτήσεις μόλις μας δοθούν, θα εκκινήσουμε απευθεία την επιχείρηση με τον καλύτερο δυνατό συντονισμό μεταξύ των εταίρων. Σε ό,τι αφορά τώρα την ιατρική εκένωση, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων, περίπου 700 μπορούμε να εκτιμήσουμε, Το πρώτο βέβαια μέλημα θα είναι να ταυτοποιήσουμε τα άτομα που χρήζουν εκένωσης, γυναίκες, παιδιά, τραυματίες. Βεβαίω πρέπει να επικεντρωθούμε και στα θύματα των βομβαρδισμών, όμω υπάρχουν και, και ε, ασθενεί χρονιών παθήσεων. Και αυτοί θα πρέπει, ε, θα πρέπει να του βγάλουμε από το χαλέπι, που δεν θα είναι εύκολο. και μετά να τους μεταφέρουμε είτε στο Χαλέπι είτε σε ένα σημείο κοντά στα τουρκικά σύνορα όπου έχουμε καταστάσεις που ελπίζουμε ότι θα είναι επαρκής. Έτσι έχει η κατάσταση προς το παρόν, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Περιμένουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την πρόσβαση και την ε, άδεια που θα μας δοθεί για να έχουμε πρόσβαση. Ελπίζουμε τουλάχιστον και από την άλλη πλευρά να κατανοήσουν το μήνυμά μας, ότι αυτή είναι μια ανθρωπιστική και μόνο επιχείρηση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί και εγώ καθυστέρησα να φτάσω. Θα μπορούσα να σας μιλήσω σε μεγαλύτερο βάθος σε ό,τι φορά την κατάσταση στα βόρεια σύνορα. Διακόπτη, Πρόεδρος. Παρακαλώ τα πηγαδάκια να μεταφερθούν εκτός της αίθουσας. Σας παρακαλώ, γιατί δεν είναι εύκολο. Ξέρω ότι έχετε πολλά να φροντίσετε, αλλά αν γίνεται να τα κάνετε αυτά εκτός. Ναι, έτσι αλλιώς ε, ολοκληρώνω. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση de facto που έχει διαμορφωθεί από τις τουρκικές αρχές. Αναφέρομαι στην ε, μεθοριακή περιοχή Σαραμπρούς που όντως ε, έχουμε μία de facto ε, ασφαλή ζώνη που δεν στηρίζεται από κάποιο ψήφισμα ή άλλη απόφαση. Η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στις ανθρωπιστικές αποστολές. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί το προσωπικό μας να έχει πρόσβαση σε αυτή τη ζώνη και ποιοι άτυποι κανόνες ισχύουν. 3.000 Σύριοι έχουν αξιοποιήσει αυτές τις εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχει βεβαιωθεί αυτό, για να περάσουν τα σύνορα και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Να, να τονίσω μόνο το εξή. Επανέρχομαι στο Χαλέπι. Πρέπει να δούμε και ποιοι θα καταστήσουν δυνατή αυτή την επιχείρηση και οι ένοπλες δυνάμεις και η αντιπολίτευση. Μεταξύ αυτών των ε, συνομιλητών είναι και η τουρκική κυβέρνηση, γιατί χρειαζόμαστε πρόσβαση σε ένα από τα μεθοριακά σύνορα και έχουν πει και το έχουν κάνει και πράξη ότι θα μας στηρίξουν ως προς την υλοποίηση της επιχείρησης. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Επίσης, μας προβληματίζει ιδίως η κατάσταση στα σύνορα με την Ιορδανία, οι εταίροι μας ε, έχουν ε, την πρόκληση ότι πρέπει με αυτό σχέδιο τρόπο ε, να παράσχουν αυτές τις βασικές υπηρεσίες σε περίπου 80.000 άτομα που αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί στα σύνορα και έχουν εγκλωβιστεί στα σύνορα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω βέβαια, γιατί θέλετε κι εσείς να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Δεν θέλω να φανώ απεσιόδοξος, όμως ε, πραγματικά τώρα έχουμε την εντύπωση ότι είναι σαν να είμαστε στα πρόφυρα μιας ε, ακόμα χειρότερης κατάστασης, χειρότερης από ποτέ. Όλα τα φανάρια πάνε στο κόκκινο, αν θέλετε. Οι χορηγοί έδωσαν τα υπεσχεμένα. Έχουμε τους πόρους λοιπόν για τους εταίρους. Το Ιράκ ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα υποχρηματοδότησης ανθρωπιστικών ε, αναγκών, αλλά ω προς τη Συρία τουλάχιστον τα χρήματα υπάρχουν τέλο πάντων. Εντάξει, βέβαια είναι ευρύτερο το ζήτημα ε, ανθρωπιστικό. Όμω το πρόβλημα δεν είναι οι πόροι, είναι η απόλυτη πολιτικοποίηση του ζητήματο. Μιλήσετε κι εσείς, ε, κυρία Πρόεδρε, για τον βομβαρδισμό του κομβόη και αυτό οδήγησε σε απόλυτη παράλυση της ανθρωπιστικής βοήθειας εάν δεν αναλυφθεί εγκαίρως και ταχύτατα δράση για να πείσουμε τους υπεύθυνους χαράξης της πολιτικής όχι για την ευημερία αλλά για τη διάσωση ζώων στη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους θα ήθελα να πω το εξή. Είπατε ότι δεν είχατε την άδεια. Ποιος είναι υπεύθυνο για την χορήγηση αυτών των αδειών και πού ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Στη Συρία, στο Ανατολικό Χαλέπι, κοντά στα σύνορα με, τη με την Ιορδανία και στην περιοχή κοντά στα σύνορα με την Τουρκία ε, θα μεταβεί κάποια ανθρωπιστική βοήθεια. Τι είναι το εμπόδιο, είναι η Συριανή κυβέρνηση, είναι οι δυνάμεις των ανταρτών, πού είναι τα εμπόδια για την ανθρωπιστική βοήθεια και γιατί δεν μπορεί να περάσει καμιά από αυτές τις περιοχές η ανθρωπιστική βοήθεια. Απάντηση. Η απάντηση είναι απλή. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση της Συρίας. το κομβόι θα αρχίσει να κινείται και θα δούμε ε, που ε, οι διάφορες δυνάμεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα πόσχουν από κάθε επιθετική πράξη έναντι της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά πόσο πραγματικά θα εκπληρώσουν αυτές τις δεσμεύσεις. Όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή και γίνονται κάποιες συζητήσεις μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και ΑΣΑΔ... Ε, ε, βεβαίως, ε, όπως σας είπα, θα ξεκινήσει το κομβόι και ICRC. Ε, και όλα αυτά ε, θα τα πω πολύ απλά. Όσο δούλευε η, ανθρωπιστική, η ομάδα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, υπήρχαν κάποια προγράμματα τα οποία, επί των οποίων γινόταν κάποια διαπραγμάτευση όσον αφορά τους, τον προορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, πότε και τους εταίρους. Και ήταν ε, προγράμματα τα οποία είχαν γίνει αποδεκτά από αυτούς που είχαν τον έλεγχο αυτής της ε, περιοχής. Και ε, πολύ συχνά υπήρχαν βέβαια κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αυτό τα παιχνίδια. Αλλά όπως σας είπα, μέχρι τότε η διαδικασία ήταν αρκετά ικανοποιητική. Ένα από τα μηνύματα τα οποία εμείς απευθύναμε προς τον κύριο Δενιστούρα και ήταν ε, πολύ προφανές ότι η ομάδα ότι θα έπρεπε να στείλουμε αυτό το μήνυμα για να κρατηθεί ζωντανή ανθρωπιστική βοήθεια. Έστω και αν ε, ε, συνδέεται με κάποιο πολιτικό εργαλείο, δεν θα πρέπει να διαλυθεί αυτή η πλατφόρμα, γιατί ε, πραγματικά είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε για να έχουμε κάποια αποτελέσματα, να παράσχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Και έχει γίνει μια συνάντηση, νομίζω ότι θα ακολουθήσει άλλη μία αυτή τη βδομάδα, αλλά εάν οι εταίροι τελικά αποκρύπτονται πίσω από πολιτικές, ε, ε, πολιτικούς διαλόγους και πολιτικά επιχειρήματα, αυτό θα, θα είναι χρήσιμο. Ε, ο κ. Γεραίρο, ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχεστε σε, αυτές, αυτή την Επιτροπή για να συζητήσετε για κάποια αφρικιαστικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, για φρικαλαιότητες, είναι αλήθεια ότι ταυτόχρονα μας δίνεται μια πολύ λεπτομερή ενημέρωση και δείχνεται μεγάλο ζήλο όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι εδώ όλοι που βρισκόμαστε εδώ συμμεριζόμαστε πραγματικά ε, τις ευχαριστίες προς τους ανθρώπους οι οποίοι ε, διαχειρίζονται την ανθρωπιστική βοήθεια και πραγματικά θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους σε πόλεις όπως το Χαλέπι και σε άλλες ζώνες. Χθες ε, είδα τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος επίσης με ενημέρωσε για την εφαρμογή της πρότασης της Αντιπροέδρου κυρίας Μοργαρίνη με δύο στόχους ε, πρωτίστως, να εγγυηθεί η πρόσβαση και η ιατρική εκένωση. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι στόχοι, όπως για παράδειγμα η παροχή ε, τροφίμων ή άλλης μορφής βοήθεια. Αλλά ε, το βασικό είναι να μπορούν να φτάσουν και το δεύτερο είναι να μπορεί να γίνει η ιατρική εκένωση, όπως επισημάνατε και εσείς. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση, γιατί όπως επισημάνατε και εσείς, η πολιτικοποίηση εκ μέρους ε, εκείνων των ε, μερών ε, των οποίων η ηγεμονική θέση διακυβεύεται εκεί είναι αυτό το οποίο πραγματικά υπονομεύει τις δυνατότητες να υπάρξει ε, ουσιαστική πρόσβαση προς τα θύματα της ε, βίας. Και από την προοπτική της ανθρωπιστικής βοήθειας, βέβαια από την άλλη, μόνο εάν πολιτικοποιήσουμε το θέμα, μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ε, έχουμε μια πρόσβαση σε εκείνους που το χρειάζονται. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια αντίφαση ότι από την άποψη της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι, αμερόληπτοι κλπ. Αλλά όταν βρισκόμαστε απέναντι σε μια σύγκρουση αυτής της μορφής θα πρέπει και εμείς να παίξουμε αναγκαστικά ένα πολιτικό ρόλο. Το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα συζήτησε ε, έκανε μια συζήτηση για την ε, Συρία, ενό ψηφίσματο για τη Συρία και είναι σαφές ότι καταδικόζουμε κάθε μορφής επίθεσης σε ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις και ανθρωπιστικούς φορείς και βεβαίως απαιτούμε την ελεύθερη πρόσβαση, αλλά φτάνουμε κάποια στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, ως πολιτικός παράγων να ε, ε, παλέψει ούτως ώστε να παίξει το πολιτικό χαρτί, ούτως ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να φτάσει εκεί που το επιθυμεί. Yeah, thank you very much. Um, um, Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Χαταλά. Πώς θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες γυναικών και κοριτσιών στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Βλέπουμε να αυξάνονται οι γάμοι με ανήλικους και έχουμε και το θέμα της σεξουαλικής βίας. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ανάγκες γυναικών και κοριτσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη. Να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται. Πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση αν αυτέ οι καταστάσεις ισχύουν. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας η οποία πραγματικά είναι σοκαριστική. Ε, Κο εδώ είναι το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να βοηθήσει, ότι έχουμε στη διάθεσή μας τα κονδύλια και ο οικονομικός παράγων στην περίπτωση αυτή δεν παίζει κανένα ρόλο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις, είναι περιορισμένοι. Και θεωρώ ότι ο Ενρική έχει δίκιο όταν λέει ότι δυστυχώς ε, είναι απαραίτητη η πολιτική διάσταση προκειμένου να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στο Χαλέπι. Γι' αυτό λυπούμε για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, μπόρεσε συσπηρωμένη να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την πολιτική της ισχύ, ούτω ώστε να αναλάβει πρωτοβουλία στο διεθνές ε, ε, τοπίο. Και έχω την, ε, το εξή ερώτημα. Αναφερθήκατε ότι υπήρξε μια ανθρωπιστική ομάδα η οποία ήταν πετυχημένη και η οποία τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα μπόρεσε να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεσματικά και η οποία πλέον δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Το ερώτημά μου έχει εξή. Ποιος ε, διαπραγματεύεται με τις ε, Ισλαμιστικές ομάδες ανταρτών στο Ανατολικό Χαλέπι. Γιατί από τη μία είπατε ότι έχετε ως δυνατότητα πρόσβαση μόνο την Συριακή κυβέρνηση, αλλά το ερώτημά μου είναι ποιος ακριβώς διαπραγματεύεται με τους Ισλαμιστές στο Ανατολικό Χαλέπι. Γιατί χωρίς τη δική του συνένεση ε, φαντάζομαι δεν θα υπάρξει πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στη Συρία είναι ένας κίνδυνος και για την ευρωπαϊκή ασφαλεία. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο, στα πρόθυρα πολέμου. Ενισχύονται οι Ρώσοι Έφεραν και πυράβλους. S300-S400 προσπαθώντας να επιβάλλουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Οι ΙΠΑ δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Γιατί θα θέσει εκείνο την κυρία Χίλαρη η κυβέρνηση του Ομπάμα και τι πιθανότητε τη για να κερδίσει τι εκλογέ. Και οι Ρώσοι έχουν πλήρη πρωτοβουλία. Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι τρομακτική. Πρέπει να καλέσουμε την κυρία Μογκερίνη και την Κομισιόν για επανάληψη των επραγματεύσεων για την ανακοχή στη Συρία. Να ζητήσουμε λοιπόν από είπα, και τη Ρωσία να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την ανακοχή και εμείς και ο ΙΕ, ο Γενικός Γραμματέας. Η κατάσταση λοιπόν είναι τρομακτική. Πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν σε παλαιότερες σειράξεις. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει μια ισχυρή θέση ότι αυτή η κατάσταση δεν γίνεται να συνεχιστεί. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να είμαστε στα όρια του πολέμου στη Συρία. και η καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους έχει πια γίνει κάτι το δευτερεύον στη Συρία. Δεν είναι το κύριο θέμα που βρίσκεται στο κέντρο της σύραξης. Αυτό είναι το μήνυμα προς εσάς στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ότι η κυρία Μογκερίνη το ταχύτερο δυνατό θα πρέπει να υιοθετήσει ισχυρή θέση κάνοντας έκκληση σε ΙΠΑ και Ρωσία να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για ανακοχή. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους συναδελφούς. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Κάποιοι πολίτες μας παρακολουθούν όλα αυτά στην τηλεόραση και έλαβα επιστολές που μιλούσαν για μεταφορές και κενώσεις ιατρικής φύσης μετά από τα κτλ για τους πιο ευάλωτους ηλικιωμένους γυναίκες, παιδιά. Τι γίνεται, γιατί τα βλέπει αυτό ο κόσμος και λέει εντάξει, εδώ πολεμάνε, αλλά οι άμαχοι που δεν εμπλέκονται, μήπως θα μπορούσαν να εκκοινωθούν εκτός από αυτούς που εκκοινώνται για ιατρικούς λόγους, γιατί έχω λάβει πολλά γράμματα, πολλές επιστολές για αυτό το θέμα. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις και για την υποστήριξη και εκτίμηση της δουλειά που κάνουμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι εταίροι μας στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ακούσαμε διάφορα σχόλια. Τα σημειώνω ως αρμόδιος. Θα τα μεταφέρω στους αδελφούς να απαντήσουν και αυτοί. Να σχολιάσω το εξής. Η σχέση μεταξύ ανθρωπιστικής βοηθείας και πολιτικής θέσης. Κάπου διάβασα τη διάταξη για την παροχή ανθρωπικής βοήθειας ως Ένωση. Υπάρχει μια αρνητή μνήμα εκεί, στη διάταξη, για τις αρχές που διέπουν την ανθρωπιστική παρέμβαση. Αμεροληψία κλπ. κλπ. Υπάρχουν όλα αυτά λοιπόν και το κάνουμε όχι επειδή θέλουμε να είμαστε καλοί, αλλά επειδή ακολουθούμε συνθήκες. Αυτές οι αρχές λοιπόν και αυτή η αντίληψη της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι το μήνυμα το ίδιο της Ένωσης. Όταν λοιπόν η Μογκερίνη η Κυριακή απόγευμα παίρνει τηλέφωνο τον Λαυρόφ και του εξηγεί τι κάνουμε και το ανακοινωθέν μα. αλλά μια πολιτική θέση και έτσι το βλέπουν και οι Ρώσοι αλλά βάσει ανθρωπιστικής παρέμβασης. Αυτή λοιπόν η ανθρωπιστική διπλωματία είναι τμήμα της διπλωματικής ατζέντας της Ένωσης. Οπότε, υπάρχει μια αμφισημία όπως λέτε, αλλά μια θετική αμφισημία. για την προστασία των πιο ευάλωτων. Συρία και γενικότερα, γιατί έχετε απόλυτα δίκιο ότι επικεντρωνόμαστε στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών, αλλά έχουμε κάνει μια τεράστια κρίση που αφορά και άλλα μέρη, μένει και Αυτή η προσέγγιση λοιπόν για τους πιο ευάλωτους και η προστασία τους βρίσκεται σε όλες τις δράσεις μας. Πάντοτε επικεντρώμαστε στους πιο ευάλωτους. Και είναι τμήμα γενικά όλων των παρεμβάσεων μας. Η προστασία λοιπόν του διεθνούς δικαίου από παραβιάσεις, τις οποίες βέβαια βλέπουμε καθημερινά, γιατί βλέπουμε ας πούμε πολιτικές εγκαταστάσεις να βορβαδίζονται και να αποτελούν στόχο. Έχουμε λοιπόν κατάφορη παραβίαση. Αλλά από τη στιγμή που θα το πούμε αυτό, αν δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής, τότε καταλήγεται σε μια κατάσταση κάπως άβολη, ένα αδιέξοδο. Να επιμείνω και πάλι ότι όλες μας, όλες μας οι παρεμβάσεις ε, καθοδηγούνται από αυτές τις αρχές. Τώρα, γι' αυτό είπατε εσείς, Πρόεδρε. Προς το παρόν, και θα είναι να το πετύχουμε, επικεντρωνόμαστε στην, στις ιατρικές εκενώσεις που αφορούν βέβαια του πιο ευάλωτους, εξορισμού δηλαδή γυναίκες και παιδιά, που είναι το αντικείμενο αυτών των εκενώσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο όλοι οι εταίροι έχουν δυνατότητα να κάνουν μια αξιολόγηση πριν, πριν αυτές οι αξιολογήσεις για το ποιοι ακριβώ θα κενωθούν. Πάντως, εξορισμού αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται σημείο και θέμα προτεραιότητας. Τώρα, νωρίτερα όταν η κατάσταση δεν ήταν τόσο άσχημη, πριν δυστυχώ πολύ καιρό που είχα πάει στη Δαμασκό, είχαμε συζητήσει ακριβώ αυτές τις τοπικές καταπαύσεις πυρός σε πολύ συγκεκριμένα μέρη που θα μας επέτρεπαν ακριβώς να κενώσουμε αυτές τις ευάλωτες ομάδες από αυτές τις περιοχές. Αλλά ούτε αυτό δεν γίνεται πια σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι η κατάσταση έχει αυθεί σοβαρά. Η συμμαχία της Συριακής Αντιπολίτευσης είπε ότι θα υποστηρίξει την εφαρμογή της κατάπαυση του πυρό και αυτών των δράσεων. Είχαμε εμείς ε, τους επαφή. Προσπαθήσαμε και μέσω αραβικού συνδέσμου να κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Και είχαμε θετικές αντιδράσεις. Τώρα όμως, για το τι συμβαίνει εκεί, εξαρτάται και από άλλους. Και ξέρετε ότι είναι και θέμα διαπραγματεύσεων και με άλλους σημαντικούς εταίρους, το ΣΑΡΚ ας πούμε. Και αυτές οι ιατρικές εκενώσεις, αν γίνουν, θα γίνουν στα γραφεία ΣΑΡΚ. Μέσω επαφών με τοπικούς εταίρους κτλ. κτλ. Ναι, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ. η Ένωση βλέπουμε ότι θα μπορούσε να δράσει αν της επιτραπεί. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε ακριβώς και την βούληση, να απολυτοσκοπήσουμε και τους άλλους εταίρους. Καταρχά, βέβαια, η Συριακή κυβέρνηση πρέπει να την έγκρισή τη και δεν είναι βέβαια αποδεκτό να είναι στόχος πολίτες. Πάντως, από ό,τι μας είπε η Επίτροπος, γίνεται πολλή δουλειά και στο παρασκήνιο. Υπόθηκε ότι θα ανοίξουν τέλο πάντων οι ανθρωπιστικές δίωδοι, αλλά ακόμα δεν το έχουν πετύχει, είναι πολύ δύσκολο. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε ότι δουλεύετε σκληρά στο παρασκήνιο και τις επόμενες μέρες ελπίζουμε να δούμε κάποια πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χειροκροτήσουμε τον ομιλητή και μη στεναχωριέστε, μη ζητάτε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εντάξει, συνάδελφοι. Ξεκίνησαμε με μια καθυστέρηση λόγω των προβλημάτων στο κτίριο, όμως ε, έχουμε ζητήσει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει έναν εκπρόσωπο για να μας μιλήσει για τον ε, τυφώνα Μάθιου ε, στην ε, Καρεβική. πιο συγκεκριμένα στην ΑΕΤ, γιατί εκεί ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα. Η Αντρόλα Καμινάρα, διευθύντρια για την ευρύτερη περιοχή, έχει έρθει εδώ. Νομίζω για πρώτη, πρώτη φορά έρχεστε στην Επιτροπή μας. Δεν έχουμε ε, ξαναβρεθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε και μάλιστα τόσο τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πριν επισέλθω ε, σε λεπτομέρειες την ανταπόκρισή μας ε, για τον τυφώνα, θα ήθελα ε, να σας δώσω μια επισκόπηση των όσων κάναμε στην ΑΕΤ τα τελευταία χρόνια και των όσων έχουμε κάνει στην περιοχή και τι θα γίνει και λόγω του τυφώνα. Υπάρχει και ένα φυλάδιο, το οποίο ενδεχομένω έχει διαμοιραστεί και στο οποίο θα φασίσω και τις ε, εξηγήσει μου. Δύο λόγια αρχικά για τα όσα κάνουμε στην ΑΕΤ τα, τελευταία, τα τελευταία χρόνια. Από το 1995 έχουμε υλοποιήσει ε, προγράμματα ανθρωπιστικά, 55 εκατομμύριων ευρώ. Περίπου 34 εκατομμύρια από αυτά αφορούσαν ε, προγράμματα με σκοπό την ε, βελτίωση της ανταπόκρισης σε ε, φυσικές καταστροφές στο νησί. Έχουμε 25 προγράμματα που ακόμα συνεχίζονται και αξιοποιούνται κυρίως για σκοπούς διατροφής και ανακούφισης τέτοιων φυσικών καταστροφών, οι συνοποιών αυτών των καταστροφών και για την αντιμετώπιση της χολέρας μετά τον ε, τυφώνα Μάθιου έχουμε αυξήσει ε, τους πόρους με 1,7 εκατομμύρια. Την Παρασκευή δόθηκε αυτό το ποσό για την αντιμετώπιση των ε, αναγκών και έχουμε κάνει μια πολύ καλή μελέτη με τους εταίρους μας επιτόπου για να δούμε τι μπορούμε να ανακατευθύνουμε στις ε, πληγήσεις περιοχές. Δεν ξέρω αν έχετε αυτό το χάρτη. Έχουμε τις δύο χερσονήσους στα ανατολικά της Αιτής. Ε, στην τελευταία σελίδα θα το βρείτε αυτό. Αυτές επλήγησαν κυρίως. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε ακόμα και όχι είναι ότι δεν υπάρχει καλή πρόσβαση σε όλες τις πληγήσει περιοχές. Και από αυτή την άποψη ε, δεν είναι πολύ ακριβή η εκτίμηση των αναγκών. Έχουμε μια εικόνα, αλλά δεν γνωρίζουμε ε, το ακριβές ε, μέγεθος του προβλήματος. Έχουμε κινητοποιήσει και ομάδες πολιτικής προστασίας, που είναι ο άλλος βραχίωνας της ΕΚΟΠ, Ήδη έχουμε μία ομάδα 10 εμπειρογνωμόνων πολιτικής προστασίας από χώρες όπως είναι η Δανία, Γαλλία, Ρουμανία, Σουηδία, που βρίσκονται επί τόπου και συμβάλλουν στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων και στην ε, επικοινωνία. Υπάρχουν προσφορές και από άλλα κρατημέλη και η Γαλλία έχει προσφέρει 65 άτομα τα οποία ήταν στη Μαρτινίκα και ε, μέλη του ιατρικού προσωπικού, όμως για να μεταφερθούν στην IT ε, πρέπει η κυβέρνηση ε, να δώσει την άδειά της. Χθε μάλιστα συναντηθήκαμε με τον πρέσβη για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε το πράσινο φως. Δεν το έχουμε λάβει ακόμα. Από το παρελθόν από άλλες εμπειρίες, ιδίως ε, μετά το σεισμό του 2010 στην ΑΕΤ, μάθαμε ότι πρέπει να αφήνουμε ε, την εκάστοτε κυβέρνηση να τίθεται επικεφαλής ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας επιτόπου. Αυτό που θέλει και η ίδια η κυβέρνηση. Αυτό έχει δημιουργήσει ορισμένες καθυστερήσεις ως προς την ανταπόκρισή μας, όμως είναι μία κοινή προσέγγιση και συμφωνούμε ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, αλλιώς ε, ενδέχεται να έχουμε προβλήματα όπως είχαμε στο παρελθόν. Όταν έχουμε πολλές ε, ΜΚΟ, πολλούς εταίρους που όλοι κάπως μαζεύονται χωρίς κανέναν συντονισμό και κάνουν ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχουν τρία επίπεδα αναγκών που πρέπει να καλυφθούν. Αυτό μας λέει και η κυβέρνηση και εδώ στις Βρυξέλλες μέσω του πρέσβη και ε, στο Πόγο το μήνυμα που έχει διαβιβάσει ο, η κυβέρνηση στον επικεφαλής της ε, αποστολής. Βασική κάλυψη αναγκών λοιπόν, ε, τροφή, στέγη, νερό. Σε ορισμένες περιοχές ουσιαστικά Όλες οι κατοικίες έχουν καταστραφεί, ιδίως στην πόλη Τζέρεμι και στην Νότια Χερσόνησο. Σχεδόν όλα τα κτίρια έχουν καταστραφεί. Ε, αυτές είναι οι άμεσες επίγουσες ε, ανάγκες. Έχουμε κάποιες πιο μεσοπρόθεσμες που αφορούν και το ζωικό κεφάλαιο, γιατί πρόκειται και για γεωργικές ε, περιοχές, με πολλούς γιοργούς και αλληλεί. Πολλές υποδομέ έχουν καταστραφεί, επομένως πρέπει να διασφαλίσουμε ε, τις ε, δουλειέ αυτών των ανθρώπων. Και βέβαια και το περιβάλλον έχει πληγεί σοβαρά, το οποίο θα λάβει πιο μακροπρόθεσμη διάσταση. Ο ΙΕ χρησιμοποιεί και την ειρηνευτική αποστολή ε, στο νησί για να αδειάσει τους δρόμους από τα μπάζα ή για να ε, ανακατασκευάσει συγκεκριμένες υποδομές και για να υπάρχει έτσι πρόσβαση και στις πληγήσεις περιοχές. Αυτά κάνουμε πάνω κάτω. Αν θέλετε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες ε, για συγκεκριμένους τομείς και περιοχές, ε, είμαι στη θέση σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, υπάρχουν ερωτήσει. Νομίζω ήταν πολύ καλή η ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν. Παρακαλώ, κυρία Θεοχάρου. Ε, εγώ θέλω να καλωσορίσω την κυρία Καμιναρά που είναι και από την πατρίδα μου και ήταν χρόνια στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Να τη συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν και να επισημάνω ότι χώρες όπως η Αϊτή μπορεί να πληγούν από ένα τυφώνα και να μην υπάρχει τρόπος προστασίας όπως, όπως συνέβη και στη Νέα Ορλεάνη για παράδειγμα ή στη Φλόριτα πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν είναι σαν ένα σεισμό όπου μπορεί να υπάρξει υποδομή προστασίας και αναφέρομαι στο παράδειγμα της Χιλής όπου ένα σεισμός 7 ρίχτερ παρόμοιος με αυτό που έγινε στην Αϊτή και την ισοπαίδωσε. Δεν είχε καμία μα καμία επίπτωση. Αν θυμάμαι καλά ήταν ένας ή δύο οι νεκροί μόνο στην ε, Χιλή σε αντίθεση με τις χιλιάδες στην Αϊτή. Ε, η Αϊτή που την γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι μια χώρα χωρίς καθόλου υποδομές όσον αφορά το δίκτυο ε, συγκοινωνιών. Οι δρόμοι για να διανύσει κανείς μια πολύ μικρή απόσταση μπορεί να χρειαστεί και τρεις και τέσσερις ώρες και οι άνθρωποι κρέμονται σαν τα τσαμπιά πάνω σε μικρά φορτηγά και μετακινούνται. Ε, με την καταστροφή της υποδομής καταλαβαίνετε ότι όλα θα πρέπει να γίνουν εξ υπαρχής. Δεν συμφωνώ με την κυρία Καμιναρά ότι η κυβέρνηση της ΑΙΤΙΣ μπορεί αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί ε, τεράστια ποσά οικονομικής ε, βοήθειας από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας θυμίσω όχι το πολύ παλιότερο παρελθόν με τον Papa και τον Baby Doc τι ζημιά είχαν κάνει όσον αφορά την ε, ηθική υπόσταση εκείνου του λαού. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Θεογάρου για τα πολύ καλά της λόγια και για το καλωσόρισμά της. Πραγματικά εκτιμώ πολύ τα όσα είπε και έχω επίγνωση του γεγονότος του πόσο καλά γνωρίζει την ΑΕΤ και σέβομαι τις απόψεις της. Όσον αφορά τις υποδομές έχετε δίκιο είναι μια χώρα όπου οι υποδομές και η πρόσβαση σε αυτές είναι ιδιαίτερος προβληματική. Γι' αυτό χτες μιλώντας ε, στα, με τα Ηνωμένα Έθνη και ε, λέγοντας ότι υπάρχει πρόσβαση στις περιοχές αυτές, ε, μου έδωσαν την πληροφορία ότι οι ρευτικές δυνάμεις ε, έχουν τέτοια προβλήματα πρόσβασης. Και, αλλά ορισμένοι από τους πολίτες έχουν κάποια εμπειρία και φροντίζουν να κατασκευάσουν τις ε, υποδομές, ε, γέφυρες κλπ. Ούτως ώστε να θέλει εξασφαλιστεί μια καλύτερη πρόσβαση εντός της ΑΕΤΙΣ. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν υποδομές ευρύτερα σε αυτό το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και το θέμα βεβαίως είναι κατά πόσο θα πρέπει να περάσουμε από την κυβέρνηση ή να δράσουμε άμεσα. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι είμαστε σε επαφή με όλους μας τους εταίρους και επιτόπου ε, και με όσους έχουν, φορείς έχουν αναλάβει το συντονισμό της ανακουφιστικής βοήθειας και από τη Νέα Υόρκη μας είπαν ότι ε, θα πρέπει να υπάρξει ως δυνατόν ε, μεγαλύτερος, περισσότερος συντονισμός μέσω των κυβερνητικών δομών, ούτως ώστε να αποφευθεί η σύγχυση και η ενεποτελεσματικότητα όσον αφορά ε, την ε, χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ταυτόχρονα έχουμε και 20 άτομα τα οποία εργάζονται εκεί επί τόπου ε, αξιολογούν τα όσα συνέβησαν αυτή τη στιγμή τύψω τυφώνα στην περιοχή αυτή. Έχουμε μια ενισχυμένη ομάδα, έχουμε μια ομάδα τεχνικής συνδρομής ε, και την ενισχύσαμε ώστε να έχουμε μια ακριβή ιδέα εν σχέση με το τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν δεν ε, είναι μόνο η κυβέρνηση αυτή η οποία μας ενημερώνει, ωστόσο συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση προκειμένου να παρασχεθεί πιο αποτελεσματικά ανθρωπιστική βοήθεια. Και ε, εσείς ξέρετε την IT και ξέρετε ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εν σχέση με το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Ε, γιατί έχει καλύτερη πρόσβαση και στις πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο. Ε, είναι οι τοπικοί φορείς πολλές φορές αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να μας ενημερώσουν και μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί μόνο εφόσον έχουμε κάποιους εταίρους ή εφόσον έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους εκεί. Άρα η εικόνα είναι κάπως μεικτή, δεν είναι άσπρο μαύρο. Έχουμε τον κύριο Ανιτσέτο από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς θα ήθελα να πω ότι στην ΤΕΦΚΟ ε, έχουμε μια στενή συνεργασία με τους συναδέλφους από την ΕΚΟ και παρακολουθούμε και το σύνεγγι στην κατάσταση. Η ΑΙΤ με διαφορετικούς όρους είναι η πιο φτωχή χώρα της περιοχής και ήδη συνεργαζόμαστε μαζί τους στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων, στο πλαίσιο ε, ε, και έχουμε ένα, χαρτοφυλάκιο 420 ε, εκατομμυρίων όσον αφορά την ε, παραδοσιακή βοήθεια προς την ΑΕΤ και μια από τις βασικές πτυχές είναι το, το δίδαγμα το οποίο αντιλήσαμε από τον προηγούμενο σεισμό. Είναι ότι θα πρέπει να συνδέσουμε την ανοικοδόμηση με την ανάπτυξη. Και αυτή είναι μια πτυχή στην οποία δίνουμε μεγάλη σημασία και επαναλαμβάνω έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την ΕΚΟ εδώ και αυτή τη βδομάδα προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να αναπροσανατολίσουμε τις παρούσες επιχειρήσεις μας ούτε ώστε να προσαρμοστούμε στις τρέχουσες δραστηριότητες να προσαρμόσουμε τις τρέχουσες δραστηριότητες στις νέες ε, προϋποθέσεις που δημιούργησε η καταστροφή του Μάθιου. Και ο, ο Γενικός μας Διευθυντής, ο κ. Μασαρβίση, έκανε, επισκέφθηκε τη χώρα, θα επισκεφθεί τη χώρα, συγγνώμη, στις 24 και 25 Οκτωβρίου, ε, με αφορμή την υπουργική συνάντηση στο Σαν Ντομίνγκο και θα πάει εκεί νωρίτερα ούτω ώστε να μπορέσει να επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές και να σχηματίσει μια άμεση εικόνα. Και όπως σας είπα αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε πώς να αναπροσανατολίσουμε τις επιχειρήσεις μας ούτως ώστε να προσαρμοστούμε στις νέες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα ε, να υπογραμμίσω πραγματικά τη στενή συνεργασία με την ΤΕΦΚΟ γιατί είναι μία από τις χώρες ε, προτεραιότητες τις οποίες έχουμε ορίσει από κοινού ούτε ώστε πραγματικά να εξετάσουμε και την εφαρμογή που γίνεται και το πώς μπορεί να λειτουργήσει η αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου. Το δεύτερο βεβαίως, αυτό το οποίο είπατε, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά προβλήματα στη χώρα. Και ε, ξέρετε ότι έχουν αναβληθεί εκλογές οι οποίες ε, πρόκειται να λάβουν χώρα την ερχόμενη Κυριακή λόγω των προβλημάτων με τον τυφών. Άρα λοιπόν ε, υπήρξαν και πολιτικές επιπτώσεις. Πρόεδρος, γιατί κάποιοι έλεγαν στο BBC ότι ο τυφώνας έπλεξε πολλές περιοχές, πολλές χώρες, αλλά στην IT το πλήγμα ήταν ισχυρότερο γιατί δεν ε, υπήρξε καμία ε, υποδομή, καμία προετοιμασία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε κάπως αργότερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει, αλλά είχαμε προβλήματα με την ασφάλεια είχαν οι προηγούμενοι ομιλητέ μας. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 16 της έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα το 2015. Ξέρετε ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στην εφαρμογή των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και εκπονείται μια γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση για την υποεποτροπή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων ε, και η συγητή μας είναι ο κύριο Πρέντα. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Θα ήθελα να παρέμβω ε, σχέση με το τελευταίο σημείο, αλλά επειδή είμαστε κάπως ε, βιαστικοί, δεν μπόρεσα να το κάνω γιατί οι εκλογές στην ΑΕΤ πραγματικά αυτά είναι μια τεράστια συζήτηση και δεν μπορώ να ξεχάσω ε, τι παρατήρησε εκεί η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε εκλογέ. Άρα πρόκειται για ένα ευαίσθητο σημείο. Τώρα θα περάσω όμως στο σημείο 16 όπως μου είπατε για να σας πω ότι και είχα τη δυνατότητα να θεωρήσω στην προηγούμενη εντολή την ε, γνωμοδότηση της Υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ήμουν και εισηγητής επίσης την περασμένη χρονιά στην Επιτροπή Δικαιωμάτων για την έκθεση αυτή. Και όλα αυτά σας λέω για να σας πω ότι έχω απόλυτη συνείδηση της συμβολής της δικής μας Επιτροπής γιατί ε, πράγματι θα ολοκληρώσει τους προβληματισμούς τους οποίους κάνουμε στην Υποπατροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση, κύριε Νόισερ, ευχαριστώ γιατί πραγματικά θα πρέπει να με ακούσετε. Η έκθεση είχε υιοθετηθεί από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου του 2016 και παρουσιάζεται σε μια πιο πυκνή μορφή από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για την συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης και ήδη αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χαιρετήσουμε, γιατί στο παρελθόν αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε. Και ε, εμεί επιμείναμε από τη δική μας πλευρά, ούτως ώστε το κεφάλαιο αυτό να εισαχθεί εδώ. Τώρα, ε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε βέβαια κατά πόσο είναι επαρκή η μισή σελίδα. Αλλά λόγω τη γενικότερης οικονομία του κειμένου, το οποίο όπω σα είπα είναι αρκετά πιο πυκνό αυτή τη φορά και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα σημαντικό θέμα. Ε, αλλά ε, στο οποίο όμως όλοι συμφωνούμε. Άρα λοιπόν ε, δεν νομίζω ότι το μήκο, η έκταση του κειμένου μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Τώρα θα πρέπει να η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει στα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχει μία σχέση μεταξύ, αλεξάρτησης μεταξύ ε, ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει μια διασύνδεση. Άρα χωρίς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εξαλείψουμε τη φτώχεια ούτε να εκπληρώσουμε τους στόχους της βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Άρα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να μπουν στην καρδιά των δράσεων που θα γίνουν. Ε, και να εισαχθούν με εγκάρσια τρόπο ε, σε όλες τις ε, πρωτοβουλίες και τους στόχους που περιλαμβάνονται σε αυτή την ατζέντα. Η Υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι δείκτες ότι ώστε να λαμβάνονται υπόψη πάνω τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρξει μια εγγύηση της ε, διαφάνειας. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να επιμείνουμε επίσης ε, και στο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης ε, αριθμός υπαριθμών 16 ούτως ώστε να τα ανθρώπινα δικαιώματα και η χρυσή διακυβέρνηση να επαγορέψουν την, τον προσανατολισμό μας. Επίσης αναφέρονται κάποιες δράσεις ούτως ώστε να συμπεριληφθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επιχειρησιακό επίπεδο στις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης. Η εργαλειοθήκη της προσέγγισης αυτής έχει ε, καταρτιστεί αλλά θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση με τους εταίρους μας και θα ήταν καλό όπως αναφέρεται στο τέλος της ετήσιας έκθεσης, να γίνει μια αξιολόγηση, να γίνεται μια αξιολόγηση της εργολεθήκης αυτής στο επίπεδο των αντιπροσωπιών, ώστε να δούμε κατά πόσο λειτουργεί καλά ή χρήση βελτιώσεων. Ε, μας χρειάζονται οι αντιδράσει τους λοιπόν και η αξιολόγησή τους, γιατί μπορούν οι αντιπροσωπίες να πούν πράγματα χρήσιμα για μας. Τώρα, από τη μία είναι προφανές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναγκαίο συστατικό του πολιτικού διαλόγου με όλους τους εταίρους των, μας των αναπτυσσόμενων χωρών. Από την άλλη, όπως είμαι, καθώς είμαι εισηγητής για τη συνεκτικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής, θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία της ε, PCD και την ανάγκη να υπάρξει ένας ε, συντονισμός μεταξύ όλων των εργαλείων της ε, προσέγγισης ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα. Ο Τέλος, υπάρχει ένα απλό μήνυμα το οποίο αφορά τη συνέχιση της ε, της των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο αναμένουν από εμά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Γιατί οι πολίτες ε, αναμένουν από εμά να κρατήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των ε, δράσεών μας. Δεν είστε μόνο εισηγητής για αυτό το θέμα, αλλά και για το επόμενο. Είναι η μέρα σας σήμερα. Φανσουλίκα, τρίζεις να το λόγο, Φανσουλίκα πρώτος. Κυρίε και κύριοι, να ευχαριστήσω καταρχά τον εισηγητή για τη σύνταξη αυτή τη πλήρου έκθεση, πιστεύω. Δυστυχώ φαίνεται να υποχωρεί η δημοκρατία σε πολλέ χώρε. και ο λαϊκισμός, ο εξαμισμός και οι παραβιάσεις δικαιωμάτων αυξάνονται, ιδιαίτερα σε χώρες όπως την Αφρία και στην, στην Ασία και στην Αφρική. Θα πρέπει να εποπτεύουμε τα θέματα αυτά και να δούμε με τι μέτρα θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σχέση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακυβέρνηση ε, ασφάλειας και εξάλληψη φτώχεια και επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Εμείς περνόμαστε στην πρώτη γραμμή προασπίση των δικαιωμάτων παγκοσμίω και θα πρέπει τα εργαλεία μας να είναι σωστά και κατάλληλα για τους πληθυσμού και τις ΜΚΟ που εργάζονται. Πρέπει λοιπόν στις εταιρικές σχέσεις ο σεβασμό η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ενθαρρύνεται και να προωθείται και όλα αυτά να γίνονται με τρόπο βέβαια αυτές οι συμφωνίες που να μην θίγουν την οικονομία της Ένωσης αλλά να προωθούν τη δημοκρατία και τους περιβαλλοντικούς κανόνες και εντός και εκτός της Ένωσης. Τώρα ιδιαίτερα που αντιμετωπίζουμε το θέμα μαζικής μετανάστευσης να δούμε τα βαθιά αίτια του φαινομένου, κυρίως η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτου δικαίου και τα θέματα ασφάλειας. Για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία, αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ω μη διαπραγματεύσιμα ως θέματα στο πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες. Μέσω της κοινωνίας των πολιτών και μέσω ΜΚΟ θα πρέπει να ασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας είναι αποτελεσματικές. Όταν πολλαπλασιάζονται οι συμφωνίες επενδυτικές, να υπενθυμίσουμε στην Κομισιόν ότι συμφωνίες με επικίνδυνες χώρες θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνουν δεσμευτικές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η Κομισιόν θα πρέπει συστηματικά να διεξαγάγει αξιολογήσεις στις συμφωνίες αυτές. Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη σχέση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης και να ζητήσουμε να δοθεί περισσότερη σημασία στο ρόλο της ανάπτυξης, συνεργασία για την ανάπτυξη στις εκθέσεις μας. Προσβλέπω στις τροπολογίες και ελπίζω να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι ώστε να στηρίξουμε και να έχουμε τελικά μια ισχυρή θέση. Και ευχαριστώ και τον συνάδελφο από τη Ρουμανία, τον κύριο Πρέντα. Σα ευχαριστώ όλου. linguistic... Ναι, λέει πρόεδρος, η πρόεδρο, Βλέπουμε το πόσο καλή είναι στι γλώσσες οι Ρουμάνοι φίλοι μα. Αγγλικά, γαλλικά. Είστε φοβεροί. Κυρία Μαρίνα Αλμπιόλ. Ευχαριστώ. Εμείς πιστεύουμε ότι η έκθεση δεν περιλαμβάνει τις κύριες προκλήσεις σχετικά με τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρωπιστικά μετά τα τελευταία χρόνια. Οπότε οι τροπολογίες μας αυτό θα αφορούν. Καταρχάς, την ανάγκη να τονίσουμε την απόρριψη οποιασδήποτε χειραγώγηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τους πρόσφυγες, να πούμε ότι αποτελούν ένα, ένα από τα κυριότερα πεδία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2015 και φέτο. Επ' αυτού θα καταθέσουμε τροπολογίες για να επενθυμίσουμε ότι το άρθρο 13 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καθορίζει την μετανάστευση ω ανθρώπινο δικαίωμα για τους πρόσφυγε, μιλάει συγγνώμη Επίση, βλέπουμε να παραβιάζονται κατάφορα και συνεχώς τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και μέσω συμφωνιών όπως συμφωνία με την Τουρκία που συστηματικά παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που επιβάλλει η αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους στις στοχές χώρες και περιορίζει τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να περιλάβουμε στην νομοδότηση τις επιπτώσεις της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες χώρες, φτωχές χώρες, που αποτελούν πύλη εισόδου για τις πολυεθνικές που πολύ συχνά διαπράττουν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι επίση σημαντικό, θεωρώ, η γνωμοδότηση να υπογραμμίζει την άμεση σχέση μεταξύ στρατιωτικών παρεμβάσεων που στηρίζονται από χώρες μέλη και την αύξηση των παραβιάσεων των άνθρωπινων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις όπως Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη και πώς αυτές οι επεμβάσεις οδήγησαν σε παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τέλος, θα υπογραμμίσουμε τη σημασία τη δικαιοσύνη παγκοσμίω για την καταπολέμηση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα εκφράσουμε τη λύπη μα για το γεγονό ότι κάποιε κυβερνήσει χωρών μελών περιορίζουν ακριβώ το εύρος αυτή τη παγκόσμια δικαιοσύνη και κατά συνέπεια περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαστών να διερευνήσουν εγκλήματα και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξαναλέω, οι τροπολογίε μα θα ακολουθήσουν αυτή την οδό και ελπίζω τέλο πάντων να κάνουμε καλή δουλειά σε συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Η κυρία αλλά ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορούμε να πούμε ότι και και η Βάιτχόσαρ και η Πρέντα εκθέσεις είναι πολύ καλές. Να διευκρινίσω μόνο τα εξή. Καταρχάς θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για τη σχέση μεταξύ Ανάπτυξη και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο είναι πολύ ευρύ και αφορά δεκάδες εκατομμύρια άτομα. Φέτο είδα ότι στην Νοτιοανατολική Ασία το φαινόμενο αυτό τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα έντονο και οδηγεί σε διακρίσεις. Για την έκθεση Vanderholzer, ίσως θα μπορούσαμε στις παραγράφους από 30 μέχρι 37, εκεί που μιλάει για πρόσφυγες, ετούντες άσυλο, μετανάστες, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για την ανάγκη των μεταναστών και αυτών που ζητούν άσυλο και να πεθυμίσουμε το ότι τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να αποκλείουν από εκεί. Και ξέρουμε ότι γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα εδώ στενός και θα πρέπει να το πεθυμίζουμε όπου μπορούμε. Τώρα για την προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην έκθεση Πρέντα νομίζω είναι καλή, είναι θετική. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να πεθυμίσουμε την Κομισιόν και στην ΥΠΑΔΙΚ εκπρόσωπο ότι θα πρέπει τουλάχιστον να δυναματίζει σωστά το ρόλο της και είναι σωστό που το αναφέρουμε εδώ. Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η έκθεση αυτή αφορά το εκκληστικό όργανο της Ένωσης. Μιλά για τα θερμα δικαιώματα, αλλά λέγεται ότι θα έπρεπε να κάνει η Ένωση συνολικά, η υπηρεσία εξωτερικής δάσης και ολόκληρη η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον να ζητάει το λόγο. Η κυρία Ρινάλντι από την Κομισιόν κάτι θα θέλει να πει. Κυρία Ρινάλδη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την ενθάρρυνση για συνέχιση της δουλειά μας και της προσέγγισής μας. Είχαμε αυτή την εργαλειοθήκη ως αρχή που υιοθετήθηκε το 2014 και τη χρησιμοποιήσαμε την εργαλειοθήκη για να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία και τώρα εκπαιδεύουμε τους συναδέλφους της για να αρχίσουν να τη χρησιμοποιούν αυτή τη μεθοδολογία. Για την επόμενη εκθέση λοιπόν, για το τι κάναμε φέτος, θα δείτε περισσότερα. Ίσως είναι νωρίς να μιλήσουμε για αξιολόγηση. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να δούμε αν είναι σωστή η βάση αυτής της συνεργασίας, γιατί πρέπει να δούμε ακριβώ τις πρακτικές των συναδέλφων και το κατά πόσο έχουν αλλάξει τέλο πάντων τις προσεγγίσεις και τι νοοτροπίε. Αλλά νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκπαιδεύουμε συναδέλφου, αλλάζουμε και τις εσωτερικέ μα διαδικασίε ώστε να διασφαλίσουμε το ότι λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο project το οποίο αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε και είμαστε διαθέσιμοι να ενημερώσουμε την Ευρωβουλή για τα βήματά μας για να εφαρμόσουμε αυτή τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέντα. Μάλιστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που μίλησαν με θετικά λόγια για την γνωμοδότηση. Θα ήθελα να διευκρινίσω, ακόμα και αν ε, ο κομμουνιστής συνάδελφος ε, απεχώρησε, είπε ότι έπρεπε να ψηφίσει σε κάποια άλλη επιτροπή. Παρά αυτά θα ήθελα εγώ να επισημάνω ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι εξαιρετικά σύντομη. Μόλις 1500 χαρακτήρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ξέρετε και, τις, και τους περιορισμούς που έχουμε όταν συντάσσουμε τα κείμενά μας. Δεν είναι λοιπόν η ετήσια έκθεση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σε 1500 χαρακτήρες λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαριθμίσουμε όλα όσα θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά και επίγοντα. Τις αμερικανικές παρεμβάσεις, ε, ε, τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, όλες αυτές τις θεματικές και προβληματικές που μας απασχολούν. Είναι λοιπόν αδύνατον να τα περιγράψουμε όλα αυτά. Είναι ο φυσικός περιορισμός που τίθεται λόγω των χαρακτήρων. Πρόκειται λοιπόν για μια γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής Ανάπτυξης, υπενθυμίζω, για την ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, που καταρτίζεται αυτή τη στιγμή θα συμπεριλαμβάνει επίσης πάρα πολλά διαφορετικά θέματα. Εδώ λοιπόν από πλευρά δική μα επιτροπή πρέπει να θίξουμε τα πλέον απαραίτητα στοιχεία ε, για την ετήσια έκθεση. Και καθώ την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήδη απίθυνα έκλεισε για να υπάρξει κάποιο συντονισμό και συνοχή στο έργο των δύο επιτροπών. για αυτό το λόγο και ελπίζω να μην θεωρηθεί ως ε, βούληση παρέμβασή μου απόψει σα. απλώ θα ήθελα να δείτε με μεγαλύτερη προσοχή την ε, έκθεση της Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί δεν πρέπει εδώ πέρα να βάλουμε στοιχεία και μετά να δούμε ότι ήδη υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Τελικά λοιπόν ε, θα επαναλάβουμε αυτά που ήδη υπάρχουν στην έκθεση. Δεν έχει νόημα αυτό. Να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια όταν υπάρχουν ήδη αυτά τα θέματα μέσα. είναι πιο εύκολο για κάποιου που είναι ήδη ε, μέλη τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμω νομίζω ότι όλα τα μέλη τη Επιτροπή ε, Ανάπτυξη μπορούν να διαβάσουν την έκθεση ε, πριν προσπαθήσουν να ανακαλύψουν και πάλι μια νέα ήπειρο. Ιδίω ο κύριος Βάντεν Χόλτσερ, ένας πολύ δεκεκριμένος συνάδελφο από τους σοσιαλιστές, είναι αυτό που έχει αναλάβει το ζήτημα. Επομένω, καλό πιο συγκεκριμένα του σοσιαλιστές να μην επαναλάβουν την ίδια προσπάθεια, γιατί πρέπει για το ίδιο, να μην έχουμε το ίδιο κείμενο δηλαδή. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέντα. Χριστιαν, προθεσμή υποβολή τροπολογιών στι 13 ε, ε, Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, έχει δίκιο. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένα μακροσκελέ κείμενο ε, για να έχουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Ναι, κάποιε φορέ είναι καλή ιδέα αυτό που αναφέρει, εκτό μικροφώνου βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι το μήνυμα να είναι σαφέ, όχι να έχουμε πολλέ τροπολογίε. Yeah, and we have another opinion. Okay, so deadline for amendments 30. Εντάξει, μέχρι τι 13 Οκτωβρίου λοιπόν στι 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο σημείο 17. Έκθεση πρωτοβουλία για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Πολύ σημαντική έκθεση. Σημαντική γιατί το να διασφαλίσουμε ότι είναι αποτελεσματικέ οι προσπάθειέ μα ε, επιτόπου και εξαλείφουν τη φτώχεια είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει όμω και μία ε, διεθνή διάσκεψη, συνάντηση υψηλού επίπεδου στην Κένια στα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεσή μας λοιπόν ε, θα συμβάλλει στις εργασίες αυτής της διάσκεψης. Ο κύριος Πρέντα είναι εισηγητής, θα μας τα εξηγήσει λοιπόν όλα αναλυτικά και θα μας αναφέρει τις συστάσεις του για το ποιες θα πρέπει να είναι οι δικές μας προτεραιότητες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αρχικά να πω ότι υπενθυμίζω ότι είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μετά τις θερινές διακοπές Λαμβάνοντα υπόψη τι παρατηρήσει των συναδέλφων, έχω καταρτήσει ένα σχέδιο έκθεσης, το οποίο έχετε λάβει. Σκοπός αυτή της ε, πρώτης ανταλλαγή απόψεων, το είχα αναφέρει και τότε, είναι να ε, διαρθρώσουμε θέση ως κοινοβούλιο πριν από την ε, διάσκεψη αυτή που θα λάβει χώρα στο Ναϊρόμπι στα τέλη της χρονιάς, όπως αναφέρατε. Θέλαμε επίσης να επηρεάσουμε την θέση της Ένωσης αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση. Ε, μία θέση που ακόμα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση ε, και με το Συμβούλιο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε προπαρασκευαστικό στάδιο ε, για την διάσκεψη του Ναϊρόμπι και θα ήθελα να αναφέρω ότι στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στη Σεούλ έλαβε χώρα η ενδέκατη συνάντηση του Steering Committee ε, που προωθεί τις διαπραγματεύσεις για αυτό το τελικό κείμενο που θα υιοθετηθεί το Δεκέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως και εκπροσωπείται σε αυτή τη Διευθυντική Επιτροπή και ε, είναι καλό να έχουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες ό,τι αφορά ε, την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε αυτή την προετοιμασία ιδίω ό,τι αφορά στο πιθανό σημείο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ήδη έχει τεθεί υπόψη των μελών ε, της ε, Διοικητικής Επιτροπής ε, η θέση μας. Αυτό λοιπόν είναι καλό για την δική μας Επιτροπή. Τώρα, επί της ουσίας της έκθεσής μου, όπως βλέπετε και στην ατολική Έκθεση, αναφέρω τα κύρια μηνύματα βάσει τριών αξώνων. Πρώτον, πρέπει να βασιστούμε στο κεκτημένο και να διατηρήσουμε ε, την ε, όθηση που υπάρχει, τη δυναμική που υπάρχει για την αποτελεσματικότητα της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. δεν πρέπει να παραλαμβάνουμε και να υπάρχουν άλλοι επικαλύψεις προσπάθειες. Και αυτό είναι σημαντικό για όλους τους εταίρους. ήδη τα έχω αναφέρει αυτά και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου για τους ε, στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, είναι να αξιοποιήσουμε καλύτερα του δημόσιου και ιδιωτικούς πόρους ε, προ όφελο τη ανάπτυξη. Η έκθεση υπογραμμίζει πιο συγκεκριμένα ότι οι τέσσερι αρχέ αποτελεσματικότητα ε, τη αναπτυξιακή βοήθεια εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν αποδείξει την αξία του σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, της, τη στήριξη προ τι αναπτυσσόμενε χώρε για να συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη από τι χώρε χορηγού. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτή την προσπάθεια, να ε, τελειοποιήσουμε ε, και να εξεργαστούμε περαιτέρω το θεματολόγιο, ε, το σχετικό, λαμβάνοντα υπόψη και τι ιδιαιτερότητε και τη διαφοροποίηση των φορέων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, όταν έχουμε πλήρη κατανόηση του ρόλου και αρμοδιοτήτων του καθένα, με διαφοροποιημένο τρόπο, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα τη ανάπτυξη. Από το θεσμικό πλαίσιο τώρα, αυτή η παγκόσμια εταιρική σχέση μετά την συνάντηση του Μπουσάν το 2011 είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τη συμπερίληψη και διαφοροποίηση της ανεπτυξιακής βοήθειας αλλά πιο γενικά θεωρώ για να προωθήσουμε μία αρμονική κατανόηση της έννοιας αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το εργαλείο. Τέλος, η τελική διακήρυξη των Ευρώπη θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να διατηρήσουμε τη δυναμική και την ε, αποτελεσματικότητα τη ανάπτυξη στο πλαίσιο του θεματολογίου 2030. Αυτό είναι η πρώτη ιδέα, το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα τώρα. Πρέπει καλύτερα να διαρθρώσουμε το παγκόσμιο οικοδόμημα η γενικότερο οικοδόμημα τη ανάπτυξη. Ήδη τα ανέφερα αυτά στο προηγούμενο μήνυμα. Μία από τα βασικά μηνύματα λοιπόν είναι ότι η Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει το ρόλο της ηγέτιδα δύναμη, που είχε λάβει και για το υιοθέτηση του θεματολογίου 2030 αλλά και για ε, την κατάρτιση του τρέχοντος ε, θεματολογίου. Η Ένωση λοιπόν θα πρέπει να συμβάλλει ε, σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση του οικοδομήματος αυτού καθώς και για την ανάληψη θέσης της ομάδας για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης. Μπορεί να έχει προσταθέμενη αξία σε σχέση με τα υπόλοιπα παγκόσμια και διεθνή φόρουμ που ασχολούνται ακριβώς με την υλοποίηση του θεματολογίου 2030. Αυτό μπορεί να γίνει εάν έχουμε δομήσει και οργανώσει σωστά ε, το ρόλο της ομάδας αυτής. Στέκομαι επίσης σε συγκεκριμένα σημεία βελτίωση, που χρήζουν βελτίωσης. Αρχικά, βελτίωση απαιτείται σε ό,τι φορά τον ε, ρόλο παρακολούθησης και την ανάληψη ευθυνών ως προς τις δεσμεύσεις. Μετά, ε, ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας και συντονισμού με αναπτυξιακούς φορείς. πέραν του όσα και με τους ε, αναδυόμενους ε, χορηγούς, την κοινωνία των πολιτών, ε, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις κτλ. Σαφής θα πρέπει να είναι και ο ρόλος της ομάδας αυτής της εταιρικής σχέσης για την αποτελεσματική ανάπτυξη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 της ε, έκθεσης για την επιτέξη των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης του 2017 και για το θεματολόγιο του 2030. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση στο πλαίσιο αυτής της διευθυντική Επιτροπής, πρόσφατα στη ΣΕΟΥ λοιπόν, ε, με ενδιαφέρουσες προτάσεις για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το θεσμικό όργανο θα ε, εξακολουθήσει να ηγείται στην όλη διαδικασία για την συνέχιση του διαλόγου, για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και της αναπτυξιακής βοήθειας ως ε, δύναμη, δύναμης για τις εταιρικέ σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτή τη ευρύτερη. Τρίτο μήνυμα. Θα πρέπει να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα και το θεματολόγιο βασικά ε, τη ε, αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη και στην Ευρώπη και ευρύτερα. Διαφάνεια του προγραμματισμού τη αναπτυξιακή συνεργασία μέσω ενό ε, πλαισίου που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχει σημαντική πρόοδος, όμως δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση από την Επιτροπή για το ψήφισμά μας το 2013, τρία χρόνια τώρα, για την κωδικοποίηση και ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών και πρακτικών στο συγκεκριμένο θέμα για να διασφαλίσουμε καλύτερη πληρωματικότητα και ε, συγκεκριμένο και αποτελεσματικό συντονισμό. Μετά υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία μπορούν να προαγάγουν περαιτέρω ε, το θεματολόγιο αυτό. νέες πρωτοβουλίες ε, τριγωνικής συνεργασίας με πιο συστηματικό και σωστό τρόπο ε, και συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, τοπικές αρχές. Μετά, σύνδεση, με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 16 και με βάση πάντα ε, στην, στο σεβασμό της κοινωνίας των πολιτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγγνώμη. Ε, πάντα πρέπει να έχουμε μια, ένα συγκεκριμένη στοχοθέτηση για την εξάλληψη της φτώχειας. Τι... Τέλο πάντων, ολοκληρώνω κάποια στιγμή. Έχω εποφεληθεί και της ε, ε, στήριξης της ε, γραμματείας. Εδώ ευχαριστώ πιο συγκεκριμένα και την Αν. λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος ήταν πιο μακροσκελές ε, του, το κείμενο. Θα ήθελα όμως κάποια ζητήματα να διευκρινίσω λόγω των πρόσφατων εξελίξεων. Ένα σημείο λοιπόν για τον ε, ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και θα πρέπει να ξαναδούμε ορισμένα τμήματα του υπό το φως των προκατακτικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 2016 που έκανε αυτή η παγκόσμια εταιρική σχέση για την αποτελεσματική ανάπτυξη που ολοκληρώθηκε μετά την δική μου υποβολή του κειμένου. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ και τη γραμματεία και πιο συγκεκριμένα την Χριστιαν ε, για τη βοήθεια που μου έδωσε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βάριν θα, μιλήσει, θα μιλήσω στα φιλανδικά, λέει ο μιλητής. Όχι, Πατρίτσια. Να ευχαριστήσω τον συγγητή για αυτή την περίπλοκη και καλή δουλειά. Κάποιες παρατηρήσεις έχω. Βλέπω ότι έχω λίγα λεπτά και θα το ξανασυζητήσουμε. Σημαντικό νομίζω ότι είναι να υπογραμμίσουμε τον στόχο που ανέφερε. Ότι πρέπει να είναι κάπως έτσι μπροστάριση Ένωση στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Έχουμε θέματα κλίματος, περιβάλλοντος κλπ. Όπου όταν είναι στην πρώτη γραμμή η Ένωση και προωθεί κάποια θέματα και κοινού ενδιαφέροντος, τότε πραγματικά πετυχαίνει σημαντικά αποτελέσματα. Αυτή η μάχη λοιπόν είναι μάχη της Ένωσης και εύχομαι να αποτελέσει θέμα και προτεραιότητας στο θεματολόγιο για την ανάπτυξη. Αυτή η μάχη δεν είναι μόνο ηθική της χρηστής διακυβέρνησης ως κάτι το οποίο επιβάλλεται και η ποιότητα. Τα αποτελέσματα και η ποιότητα των αποτελεσμάτων. Δεν αρκεί κανείς μόνο να δρά, αλλά να δει τι γίνεται με αυτές τις δράσεις στα πλαίσια του θεματολογίου 2030, ανθρώπινα δικαιώματα, βιωσιμότητα κλπ. Νομίζω ότι όμως θα έχουμε να κάνουμε όλο και περισσότερο και με άλλα ζητήματα οικονομικού χαρακτήρα που αφορά πόρους και ποσοστώσεις σε κάποιες χώρες. Ακούσαν προηγουμένως να γίνεται λόγος για την IT. Εγώ μόλις επέστρεψα από μια συνάντηση με επισκόπους από τη Συρία. Μας είπαν για τις τεράστιες ανάγκες και την καταστροφή σε διάφορες πόλεις και βλέπουμε να υπάρχει κάποια ανάγκη σοβαρή. Οπότε αυτό είναι απαραίτητο που κάνουμε. Να διευκρινίσω όμως κάποια πράγματα. Καταρχάς θα ήθελα να σε παρακαλέσω να υπογραμμίσεις και να διερευνήσει το εξή. Εντάξει, είναι σημαντικό να προωθήσουμε εσωτερικέ σχέσει και να έχουμε έτσι μια σφαιρική παγκόσμια εικόνα με μια προσέγγιση για τη δημιουργία αυτής της ομάδας που δημιουργήθηκε σε ψηλό επίπεδο, που προσθέτει τα ήδη υπάρχοντα φόρα. Όμως να προσέχουμε, να μην περιπλέξουμε υπερβολικά τα πράγματα με τη διακυβέρνηση. Τι σημαίνει διακυβέρνηση. Σημαίνει ότι εδώ έχουμε αυξημένες ευθύνε όλων όσων εμπλέκονται. Αλλά κοιτάξτε τελικά, το να πήγε κανείς σε συναντήσεις σεμινάρια, διασκέψεις. Φεύγει ο χρόνος και δεν μας μενεί καθόλου. Γιατί πολλές φορές αυτές οι σωστές έτσι δομές γίνονται αυτοαναφορικές, γιγαντώνονται και παραβλέπουμε τον στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Οπότε εγώ θα λέγα να ήμασταν έτσι προσεκτικοί σε σχέση με αυτά τα monitoring, τις εκθέσεις κτλ. Ωραία, να κράτσουμε μόνο την ουσία για την διακυβέρνηση. Το ίδιο και για την ποιότητα των πόρων και την αποτελεσματικότητά τους. Είπες κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που συμμερίζομαι. Να πω και το εξή. Κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε θαραλέα και σε αυτή την έκθεση και θα καταθέσω τροπολογία είναι το εξή. Εμεί στου διεθνεί οργανισμού θα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ κόστου λειτουργία και κόστου που σχετίζεται με τα αποτελέσματα που δημιουργούνται. Γιατί αν έχουμε 70% κόστος λειτουργίας κάποιων υπηρεσιών του ΟΗΕ, τότε κάτι πάει καλά. Δεν γίνεται να πληρώνεις 70% για το κόστος λειτουργίας και να έχει αποτελέσμα με 30%. Τα λέω έτσι ομά, αλλά περί αυτού πρόκειται. Είναι κρίσιμο αυτό το ζήτημα. Οπότε πρέπει να έχουμε το θάρρος να το θίξουμε αυτό. Γιατί μετά τι γίνεται, βλέπουμε ότι σε διάφορα μέρη στον κόσμο. Έχουμε διάφορες υπηρεσίες Επίσης έχουμε έχουν διαφορετικές περιγραφές σε σχέση με την τοπική αγορά. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο στα κόστη λειτουργίας. Αν εγώ λοιπόν δημιουργήσω μια διεθνή δομή, κοινοτική δομή, δεν ξέρω, οτιδήποτε, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε καλά τη σχέση μεταξύ κόστου λειτουργία και κόστου που αφορά το αποτέλεσμα. Αλλιώ η λειτουργία του δεν θα είναι αποτελεσματική. Τα νέα στοιχεία που ανέφερε είναι σημαντικά. Ενίσχυση των πρωτοβουλειών σε σχέση με διαφάνεια των ενισχύσεων και την εργαλεία. Το εργαλείο που διασφαλίζει τις τριγωνικές συνεργασίες, Αναπτυσσόμενε, μεσουσοδήματο, χώρε κλπ. Αυτό θα μπορούσε να διερευνηθεί με νέε μορφέ λειτουργία μαζί με αυτά που είπε ο εισηγητή. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα επαναλάβω, τα οποία έχω σημειώσει όμως εδώ και τα οποία αφορούν τέλο πάντων του κύριου πυλώνες και την προσέγγιση που ακολουθεί. Ξαναλέω, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το περιεχόμενο, πολύ αυστηρή δουλειά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αλλά να είμαστε οι πιο αυστηροί κριτέ του εαυτού μα, αν τα κάνουμε λοιπόν όλα αυτά και αν επιμείνουμε όπως λες και εσύ ώστε να είναι μπροστά η Ένωση σε αυτή τη μάχη καταρχάς στο εσωτερικό της και μετά προς τα έξω τότε νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ χρήσιμη δουλειά για την συνεργασία και το μέλλον της και για το θεματολόγιο 2030. Thank you, thank you. Ευχαριστούμε πολύ Πατρίτσια. Ο Πάβελ. Ναι, θα μιλήσω στα φιλανδικά. Aloitan protestoimalla sitä, että tuolla äskeisessä yhteiskokouksessa ei... Λοιπόν, ε, θα, ε, παραπονέθηκα ότι στην κοινή συνείδηση προηγουμένως δεν είχαμε φιλανδική διερμηνία. Εγώ γνωρίζω ότι ασφαλώς οι φιλανδοί διερμηνείς θα είχαν έρθει εάν είχαν ε, κληθεί. Και ε, στην ΑΦΕΤ επίσης δεν έχουμε φιλανδική διερμηνία παρόλο που υπάρχουν εκεί μέλη Φιλανδοί στην Επιτροπή αυτή. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε διερμηνία στα φιλανδικά. Λοιπόν, τα όσα είπε ο κύριος Πρέντα βρίσκω ότι είναι πολύ καλά είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους αποτελεσματικά γιατί είναι περιορισμένοι. Και αυτό αφορά τόσο τη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση. Σημαντικό είναι επίσης να πετύχουμε το στόχο του 0,7 και εφόσον εργαστούμε αποτελεσματικά μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Έχω μία φιλοσοφική ερώτηση, θα έλεγα, γιατί έγινε λόγος για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και τώρα μιλάμε για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Άρα λοιπόν με τον τρόπο αυτό τονίζεται ε, αυτή η εξίσωση. Δηλαδή δεν γίνεται πλέον λόγος για δωρητές και λύπτες, αλλά εξισώνονται. Ε, τώρα, όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, βεβαίως χρειάζονται εδώ πολλά εργαλεία. Και το ερώτημά μου έχει ως εξής. Θα πρέπει ίσως στην γνωμοδότηση αυτή να σκεφτούμε το ρόλο της αναπτυξιακής συνεργασίας και όσον αφορά την ε, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε εκείνες τις χώρες όπου υπάρχει μία οικονομική ανάπτυξη και υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί και ε, εάν επενδύσουμε τα χρήματά μας ε, για παράδειγμα στο Aid for Trade ε, βεβαίως ε, αυτό θα είναι πολύ αποτελεσματικό εάν δούμε το σύνολο της αναπτυξιακής πολιτικής και τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής. Και δεύτερον, εάν με τα κονδύλια αυτά ε, μπορέσουμε να παράσχουμε κίνητρα για την ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της φτώχειας και θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους ε, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προβληματιστούμε σε σχέση με τις ε, έννοιες και την ε, αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής και όχι μόνο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Και σε αυτή τη γνωμοδότηση υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αλλά ίσως θα έπρεπε να οριστεί αυτό με μεγαλύτερη σαφήνεια και ίσως θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε από κοινού. Σας ευχαριστώ θερμά. Um, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Η Χάιντι Χάουταλα. Ναι, μια και έχετε τα ακουστικά, κρατήστε τα. Και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο, ο οποίος ε, έχει δίκιο, γιατί βρισκόμαστε πραγματικά σε μια, μπροστά από μια έννοια στρατηγική σημασία. Μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική και είναι σημαντικό να το δούμε, να τη δούμε την έννοια αυτή σχέση με την αποτελεσματικότητα, αλλά τέτοιου είδου ενοιολογικέ ε, αλλαγές ε, μπορούν να γίνουν αργότερα. Αυτή τη στιγμή ε, έχει λάβει χώρα η ανάπτυξη Γι' αυτό θεωρώ ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Πρέτα είναι αρκετά πλατιά και καλή. Ε, εάν ε, δούμε τι έγινε ε, σε ορισμένες χώρες όπου οι πολίτες ήταν απογοητευμένοι γιατί δεν είχαν ε, συμπεριληφθεί η ΜΚΟ και δεν είχαν αρκετό περιθώριο ανάληψης δράσης. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε ε, περισσότερα δημοκρατικά στοιχεία εδώ. Νομίζω ότι η έννοια της δημοκρατικότητας εδώ θα είχε μία θέση. Στο σημείο 4 αναφέρονται οι διάφοροι παράγοντες, η κοινωνία των πολιτών, η κυβέρνηση, οι ιδιώτες, ο ιδιωτικό τομέας και θεωρώ ότι εδώ απουσιάζει μια ομάδα οι ερευνητές γιατί πραγματικά αυτοί έχουν μεγάλη σημασία όταν δημιουργούνται διάφορες ε, γραμμές προπολογισμού και λαμβάνονται αποφάσεις για την αναπτυξιακή πολιτική και την αναπτυξιακή συνεργασία. Και θεωρώ ότι θα ήταν σωστό να προσθεθεί εδώ αυτό το στοιχείο. Όσον αφορά το σημείο 13, εδώ θα ήθελα να αναφερθεί και η ευθύνη των επιχειρηματιών, γιατί ο στόχος είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ή δυνατόν τον ιδιωτικό τομέα. Η διασύνδεση η οποία απουσιάζει από αυτή την αλυσίδα σκέψεων είναι το ότι βεβαίως δεν είναι αδιάφορο το πώς ε, ε, επενδύονται τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα ε, και δεν θέλουμε τα δημόσια κονδύλια να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα παρά μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και μια από αυτές είναι και η, επιχειρηματική, η ευθύνη των επιχειρηματιών. Και πραγματικά αναμένω η Επιτροπή να παρουσιάσει το πρόγραμμα Responsible Business γιατί καθυστερεί η πρόταση αυτή χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους. Και θεωρώ ότι εδώ στο σημείο 17 είναι αλήθεια ότι η σημασία της αναπτυξιακής ε, βοήθειας ε, είναι πραγματικά αξιοσημείωτη στις ε, ελάχιστα αναπτυσσόμενες χώρες και μέσω αυτής μπορούν να ενεργοποιηθούν πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, εδώ εντάσσονται και πόροι του ιδιωτικού, για τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά βεβαίως προσπαθούμε να πετύχουμε το 0,7 του ΑΕΠ και να το κρατήσουν αυτό οι χώρες. Και αυτό ε, με οδηγεί στην εξή σκέψη όσον τη δικασία της Μποζάν και τη σχέση με τον ε, ΟΣΑ και τι θα πρέπει εδώ να ενισχυθεί ε, την Επιτροπή ΝΤΑΚ του ΩΣΑ. Πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή ΝΤΑΚ του ΩΣΑ θα πρέπει να είναι το κατάλληλο όργανο το οποίο να φροντίσει πραγματικά να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και να είναι υπεύθυνο για μια πιο αποτελεσματική συνεργασία. Και εδώ στο σημείο 17 αναφέρεται ότι ο συντονισμός δεν είναι αρκετά καλός και ίσως θα έπρεπε να γίνει εδώ κάτι και δεν μπορώ παρά να το υπογραμμίσω αυτό. Και τώρα που πλησιάζει και η συνεδρίαση στον Αϊρόμπι, θα ήθελα να πω στον κύριο Πρέντα ότι θα μπορούσε και εκεί να εκπροσωπηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί πραγματικά θα ήταν ανήκουστο να μην υπάρξει εκεί εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές, αλλά έχουμε Σαντάλ που είναι επικεφαλής του τμήματος της μονά που αντικαθιστά τον διευθυντή σου. Αν έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Νταν Πρέντα ε, για το έργο του και το κείμενό του. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και όντω το έχουμε και εμεί ε, διαβιβάσει στην Διευθυντική Επιτροπή του GBTC και ε, το έχουμε δώσει και σε όλα τα κράτη-μέλη. Να επανέλθω μόνο σε, στη δική μας θέση σε ό,τι αφορά ε, το θεματολόγιο και την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης. Έχουμε φύγει πλέον από το αποκλειστικό σημείο εστίασης την ανάπτυξη, την, ε, την συνδρομή μάλλον, την αρρωγή. Ε, είναι περισσότερο πλέον οι φορείς με μεγαλύτερη έμφαση στην συνεργασία για την ανάπτυξη και έτσι θέλουμε να μείνει. Νομίζουμε ότι συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση του θεματολογίου 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της ε, θέλουμε να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις τέσσερις αρχές της ε, δημοκρατικής ιδιοποίησης, ε, της διαφάνειας και της λογοδοσίας που μπορείτε να βρείτε στο GPTC. Έχουμε λάβει και μία πρόταση από το Μεξικό για μία πέμπτη αρχή να μην μένει κανένας πίσω την εξετάζουμε αυτή τη στιγμή με όλα τα κρατημέλη. Θέλουμε να αναλύσουμε πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί. Όμως ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας έχουν στείλει. Η αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες ε, τις ε, ροές αναπτυξιακής βοήθειας για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και αυτές οι αρχές θα πρέπει να ισχύουν και για τον ιδιωτικό τομέα και τις σχετικές εμπορικές ροές καθώς και την ε, συνεργασία νότου-νότου, ε, ανάμεικτες μορφές ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα και σχετικής χρηματοδότησης. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται καλό θα ήταν, αν υπάρχει δυνατότητα με τον περιορισμό που έχετε ε, στους χαρακτήρες, να αναφέρετε τα μέσα υλοποίησης άντις πλέον ε, τον SDG 17, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Θα στηρίξουμε και μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Ενδέχεται να έχετε δει το πιο επικαιροποιημένο κείμενο αποτελεσμάτων το οποίο αρχίζει να προτείνει αυτή την διαφοροποιημένη ε, στάση για να συνεχίσουμε εμείς με τις δεσμεύσεις μας, αλλά να προσπαθήσουμε να φέρουμε και να προσελκύσουμε άλλα υπάρχουν μέρη με, με πιο συγκεκριμένες ε, δεσμεύσεις. Καλό θα ήταν να το στηρίξετε κι εσείς, θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας. Θεωρούμε σημαντικό να επισημάνουμε την τριγωνική συνεργασία, αλλά θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι η συνεργασία νότου-νότου και θα πρέπει να τονιστεί περαιτέρω στην έκθεσή σας. Ένα συναδελφό σας ανέφερε ότι θα πρέπει να περάσουμε στην υλοποίηση. Ε, ο κοινό προγραμματισμό είναι η διέξοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω και αυτό καλό θα ήταν να τονιστεί περαιτέρω για να μα βοηθήσει και μας να μα δώσει μια μικρή όθηση. Αυτό είναι ένα τρόπο εμείς να υλοποιήσουμε τις αρχές της ε, αποτελεσματικότητας. Αυτά είναι συντομία, εν είδη σχολείων για την έκθεσή σας. Βεβαίως, ε, μεταχωράς μπορούμε να έρθουμε και να σας ενημερώσουμε ε, για τις συστηματικές, μάλλον στο πλαίσιο των συστηματικών ανταλλαγών απόψεων που έχουμε και με το Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, αλλά και ε, στον αερόμπι. Θα τα πούμε όλα αυτά. Δύο λόγια τώρα για την ε, Διευθυντική αυτή επιτροπή. Δεν ήμουν παρούσα, όμως και ο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή με τα χαρά θα έρθει και θα σα ενημερώσει περαιτέρω για τα όσα συνέβησαν, γιατί αυτό μα εκπροσώπησε. Πήγε πολύ καλύτερα αυτή η συνάντηση από ό,τι προηγούμενε. Ήταν πολύ πιο αισιόδοξο. Έχουμε λάβει το έγγραφο, ένα μακροσκελέστατο έγγραφο αποτελεσμάτων. Έχει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, έχει και θετικές διατυπώσεις, και, ε, όμως ε, απέχει και από κάποια άλλα σημεία. Ε, επαναλαμβάνει κάποια τμήματα προηγούμενων κειμένων τα οποία μπορούμε να αφήσουμε εκτός. Έχουμε ζητήσει εμείς κάποια επιπλέον σχόλια. Έχουμε μέχρι τις 23 Οκτωβρίου για να λάβουμε τέτοια γραπτά σχόλια. Τα έχουμε ζητήσει από όλα τα κρατημέλη. Αν έχετε και εσείς σχόλια, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να έχουμε ένα ενιοποιημένο κείμενο ε, το οποίο να μπορούμε να στείλουμε στην ε, ε, Διευθυντική αυτή Επιτροπή στο πλαίσιο των διπλωματέσεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Όμως καλύτερα θα ήταν να έρθει ο Κλάους να σας ενημερώσει γιατί εγώ δεν ήμουν παρούσα. Προετοιμάζουμε και την ε, Ολομέλεια και τη διασύνδεσή της με την GPTC για να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε την υλοποίηση των ε, στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε και κάποιες παράπλευρες εκδηλώσεις και για τον κοινό προγραμματισμό μεταξύ άλλων και θα συμμετάσχουμε και στην συνάντηση για ε, την κινητοποίηση εσωτερική χρηματοδότηση. Θα σας δώσουμε όμως και άλλες πληροφορίες σε περαιτέρω συζητήσει. Έιντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία ερώτηση. Ο κοινό προγραμματισμό είναι ένα από τα κύρια σημαία και εργαλεία αποτελεσματικότητας θεωρητικά. Όμως δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό τον κλάδο. Από ό,τι ξέρω εγώ, μόνο μικρός αριθμός κρατών μελών είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν αυτή την οδό, γιατί θεωρούν ότι θα περιοριστεί ε, η ορατότητά του. Τι συμβαίνει λοιπόν, έχουμε σαφή δεδομένα. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια αξιολόγηση για τον κοινό προγραμματισμό. Είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα πριν από μερικέ εβδομάδε, όταν είχαμε ένα τεχνικό σεμινάριο. Οι συνάδελφοί μα εξετάζουν την τελική έκθεση αυτή τη στιγμή, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί μα δείχνει ότι εκεί που νομίζαμε ότι θα περιοριζόταν ο όγκος, ε, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις, αλλά οι χώρες που επιλέγουν τον κοινό πραγματισμό βλέπουν ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ χρήσιμα. Ε, έτσι επικεντρώνεται και ο συντονισμός μας γύρω από ένα κείμενο και έτσι είμαστε πολύ πιο συνεπείς και στην πολιτική μας και στον πολιτικό μας διάλογο. Δεν περιορίζεται ο κατακαιρματισμός όσο θα το θέλαμε. Δεν βλέπουμε ότι συγκεντρωνόμαστε όσο θα θέλαμε σε συγκεκριμένο αριθμό κλάδων. Όμως βελτιώνονται τα αποτελέσματά μας και ο αντίκτυπος που έχουμε και δεν συμβαίνει αυτό που φοβόντουσαν τα κρατη να περιορίζεται η ορατότητά τους ή η δυνατότητα ε, να μιλούν με τους εθνικούς τους συνομιλητές. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με αυτή την αξιολόγηση θα διασκεδάσουμε ανησυχίες κρατών μελών που ανησυχούσαν λίγο για τον κοινό πραγματισμό. Όταν δώσαμε την πρώτη προκατακτική ενημέρωση, πρώτη φορά υπήρχε τέτοια αθρώα προσέλευση όταν θα έχουμε και τις συστάσεις και την τελική έκθεση, με τα χαράς να έρθουμε και εδώ να σας ενημερώσουμε για να ξέρετε και εσείς τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί προφανώς και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Θέλετε να επανέλθετε. Ναι, θα είμαι σύντομο. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μετά από αυτά που ακούσαμε, να ευχαριστήσω και του συναδέλφους που πήραν το λόγο. Τώρα, για την κυρία Τόγια, που χρειάστηκε να φύγει να πάει σε άλλη συνάντηση, πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις της για την ανάγκη έμφαση στην ποιότητα των αποτελεσμάτων και να αποφύγουμε καταστάσεις όπου το κόστος λειτουργίας είναι 70% και η παραγωγή αποτελεσμάτων είναι υποδεέστερη του κόστους λειτουργίας. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέει για το ότι τα πράγματα δεν πρέπει να τα περιπλέκουμε και ότι χρειάζονται δομές δομές διευκολυντικές και οι εταιρικέ σχέσεις εξάλλου αυτό βασίζονται σε αυτή την ιδέα. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Παγκόσμια προσέγγιση με τοπική εστίαση αναχώρα. Αυτό λέει το, το πλαίσιο εταιρική συνεργασία. Γι' αυτό που είπε τώρα ο κ. Βάρινεν, για το φιλοσοφικό ερώτημα που έθεσε. Έχουμε και τις προηγούμενες εκθέσεις μας και όπως είπε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν το θέμα της συνεργασίας για την ανάπτυξη αφορά αυτά ακριβώς που είπε και ο συνάδελφος. Τώρα βρισκόμαστε βέβαια στα πλαίσια μιας νέας φιλοσοφίας συνεργασία για την ανάπτυξη. Οπότε εδώ έχουμε ένα κοινό σημείο πέραν δηλαδή πολιτικών διαφορών. Η ομάδα μας αποδέχεται αυτή την προοπτική πάντως. Να ευχαριστήσω και την κυρία Χάουταλα για την έτσι προσεκτική ανάγνωση που έκανε και για τις παρατηρήσεις για την παράγραφο 13. Να πω ότι ίσως οφείλεται σε μια μετάφραση η οποία δεν είναι και τόσο ακριβής. Εκεί που μιλάω δηλαδή για την κοινωνική υπευθυνότητα, συγγνώμη, εταιρική υπευθυνότητα. Ίσως εκεί να υπήρχε κάποια παρανόηση. Μετά για τις μη μη, Εγώ θεωρώ ότι η ΜΚΟ είναι αρκετά παρούσες, αρκετά ενεργείς. Ήδη είχαμε αρκετές επαφές με ΜΚΟ και θα πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι η ΜΚΟ, εντάξει, επιθυμούν περισσότερα. Και εγώ ίδιος εργαστήκα σε ΜΚΟ και σε άλλες αντίστοιχες οργανώσεις. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους, να λένε ότι θέλουν όλο και πιο πολλά. Όμως εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι η ΜΚΟ είναι παρούσες και στην Επιτροπή μας, έτσι. Δεν είναι ότι εμείς ε, παρακούσαμε ή παραβλέψαμε αυτό που λένε ΜΚΟ για, τις, ε, για τη θεματική μας. Είναι πιο ενεργής και από κάποια μέλη μας η ΜΚΟ. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ. Ε, thank you very... Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Τροπολογίες 17 Δευτέρα του Οκτώβρη μεσημέρι. Σαντάλ, νομίζω ότι αν θέλει να καθέσει ο κόσμος τροπολογίες, να το κάνει τώρα. Ωραία, συνάδελφοι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κομισιόν. Σήμερα 18 δεν έχουμε ερωτήσεις. Σήμερα 19 διάφορα. Μήπως έχετε κάτι στα διάφορα, κάτω που δεν έχει αναφερθεί ήδη. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. 20. Επόμενη συνάντηση, 7 Νοέμβρη, στις 3. Και 8 Νοέμβρη, 9 ώρα το πρωί. Και 3 το απόγευμα. Έχουμε κοινέ συνεδρίες αύριο, συνάδελφοι. Θα σας ενημερώσουμε για την εφεπία με την Επιτροπή Δικαιωμάτων αύριο το πρωί 9, αύριο το απόγευμα για τη διατροφή. έχουμε και προσκλήσεις για ίντε και budget πέμπτη πρωί. Θα σε ενημερώσουμε πάντως. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Δερμής και Δερμής ευχαριστώ την Πρόεδρο. Έχουμε στις 5.30 τώρα τους συντονιστές. Αν θέλετε και είστε έτοιμοι να αρχίσουμε και νωρίτερα. Πάντως ευχαριστώ άλλη. γεια σας.